Κυρίες και κύριοι, περνάμε στις ε, αιτιολογήσεις ψήφου και αρχίζουμε με την έκθεση ΤΑΙΝ, πρωτόκολλο σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Ζανίτση έχει το λόγο. Λόγω των διαρκών αυξήσεων των εκρεμών υποθέσεων, το δικαστήριο για να αντιμετωπίσει το φόρτο εργασία ζήτησε να έχει ένα αυξημένο αριθμό δικαστών. Παρόλε τι προσπάθειε που κατεβλήθησαν, δεν μπόρεσε να επιτευχθεί αυτό εξέφρασα τη θετική ψήφο μου στο κείμενο της συναδέλφου η οποία αυξάνει τον αριθμό του δικαστών κατά 12 με αυτόν τον τρόπο περνούν από τους 27 στους 39. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Σάνεκ, ο επόμενος Thank you, Mr. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό γιατί έχασα τα γυαλιά μου. Να επαναλάβω ένα κλισέ. Όταν καθυστερεί η δικαιοσύνη είναι σαν να μην απονέμεται. Το γεγονός ότι παρόλη την αύξηση που άρχισε στον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων, ε, τον υποθέσεων αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων αυξάνεται κάθε χρόνο. Και νέες υποθέσεις εμφανίζονται Βεβαίω είμαι υπέρ τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να μα απασχολήσει ο φόρτο δικαστικών υποθέσεων. Οι διαρθρωτικές αλλαγές περιορίζουν τις αρμοδιότητες του δικαστηρίου. καθώς και των πενταμελών δικαστηρίων. Είμαι σαφώς υπέρ του εφηγρεμιστούν αυτές οι διαδικασίες έτσι ώστε να έχουν καλύτερη απονομή δικαιοσύνης οι συμπολίτε μου. Mr. Daniel. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Ευχαριστώ. Κατά το 18ο αιώνα ο ε, επίσκοπος Worsley του Winchester είπε ότι αυτός ο οποίος ε, ε, αναφέρεται στο νόμο δεν είναι και αυτός που τον έχει γράψει, που τον έχει συντάξει. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς ε, το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να λειτουργήσει. Είχαμε να κάνουμε με δύο φαινόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου δεν έχουν δικάσει στη χώρα του, στη χώρα από την οποία προέρχονται. Οι περισσότεροι ε, απλώς είναι πολιτικοί και μάλιστα φεντεραλιστές. Επίσης, ως προς την ε, περιγραφή των καθηκόντων βλέπουμε ότι οι αφορά θέματα τα οποία είναι καθαρά διακυβερνητικά. Δηλαδή δεν πρόκειται για δικαστές για μια συγκεκριμένη ε, αποστολή. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποφαίνεται το δέξτε σε καθαρά προδικαστικά ερωτήματα. Αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημοσίας Διοίκησης, επόμενη έκθεση. Η κυρία Τζανίκη και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης απαρτίζεται από 7 δικαστές. Η λειτουργία του όμως μπορεί να φυγεί στην περίπτωση κατά την οποία ένα από τα μέλη του ασθενεί ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για ένα εκτενέσει χρονικό διάστημα. Για να αποφύγουμε το δικαστήριο να βρεθεί, βρεθεί σε μια κατάσταση έτσι ώστε να μην μπορεί να ασκήσει το δικαστικό του έργο, το, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπέβαλε μία πρόταση κανονισμού η οποία επιτρέπει σε περίπτωση ανάγκη το διορισμό δικαστών, ε, αναπληρωτών δικαστών. Γι' αυτό το λόγο είμαι πεπισμένη ότι μία τέτοια πρόταση είναι μία λογική λύση σε ένα πρακτικό πρόβλημα που θα μπορούσε να δημιουργήσει προσκόμματα στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Γι' αυτό ψηφίζω υπέρα. Όπως είπα, κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ λογική αυτή η πρόταση λαμβάνοντας υπόψη τον διαρκώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας. Δεν υπάρχουν εφαρμόσιμες διαδικασίες για, το δικαστήριο, για την αντικατάσταση ενός δικαστή του, του Δικαστηρίου Δημόσιας Δίκησης σε περίπτωση ασθενείας. Εγώ ήμουν η υπέρ του να υπάρξει ένα ξεχωριστό δικαστήριο. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να πω ότι χρειαζόμαστε περισσότερα εξειδικευμένα δικαστήρια τα οποία θα παρέχουν εξακτομικευμένες ε, λύσεις. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε τον δικαστικό ακτιβισμό, όπου οι δικαστές προσπαθούν να αντικαταστήσουν τους εκλεγμένους πολιτικούς. Περνάμε σε ένα άλλο σημείο της ημερησίας διάταξης. Έκθεση Γκόραν Φάρμα. Η οικονομική ενίσχυση στις διευρωπαϊκές διαφορές και τα ενεργειακά δίκτυα. Czy poseł Zemke jest na sali? There is no uh, Mr. Zemke Um, at the plenary, so... Ο συνάδελφος δεν ε, είναι στο σώμα, δεν παρευρίσκεται, κυρία Τζανίκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να εκφράσει το δυναμικό του δίχως να υπάρχουν σύγχρονες και αποτελεσματικές υποδομές. Χάρη στην πρόσφαση ε, συμφωνία που επετεύχθη πριν από λίγο θα μπορέσουμε να δώσουμε μία όθηση στις επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφοριών και επικοινωνιών. Για το λόγο αυτό στηρίζω το κείμενο της συναδέλφου Φάτα, διότι πιστεύω ότι η επίτευξη νέων υποδομών θα μπορούσε θετικά να συμβάλλει στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επόμενη ε, ομιλήτρια, η κυρία Είναι πολύ σημαντικό το ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και επικοινωνιών. Αυτά είναι σημαντικά θέματα για το πρόγραμμα 2020 Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ανάπτυξη. Η χρηματοδότηση καλύπτει μόνο το 1 δέκατο των αναγκών. Πιστεύω ότι μια κοινή χρηματοδότηση θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια ασφάλεια στην παροχή ηρεκτικού ρεύματος καθώς και ανανεώσιμες πηγές. Αυτές είναι επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Τάνοκ, δεν ξέρω κατά πόσο χρειαζόμαστε ένα αναπτυξιακό σχέδιο μετά από την αποτυχία της ατζέντα της Λισαβόνας. Δεν ξέρω κατά πόσο ε, οι ομολογίες έργου θα μπορέσουν να επιλύσουν τα προβλήματά μας. Γι' αυτό θα πρέπει να αξιολογήσουμε την πιλωτική φάση, όπως είπε η ομάδα μου. Δεν χρειάζεται χρειαζόμαστε μία ε, αναπτυξιακή πορεία τύπου Keynes για το νότο της Ευρώπης. Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κόψουν τη γραφειοκρατία, γι' αυτό θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σχέδιο ευημερία. Θα πρέπει όμως να υποστηρίξουμε τις υποδομές και αυτή η πρωτοβουλία ίσως επιτύχει εν μέρη Γι' αυτό θα πρέπει να μπορέσουμε να λάβουμε αποφάσεις κατά πόσο μπορεί να προθεθεί αυτό το σχέδιο. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να πω κάτι για τα ομόλογα έργου που είναι μια δυνατότητα χρηματοδότησης έργων ε, σε ευρύτερη βάση με τη συμμετοχή ιδιωτών αλλά δεν πρόκειται βέβαια για ε, άπειρη διάθεση ε, χρηματοοικονομικών κεφαλαίων. Άρα τα έργα θα πρέπει να είναι ε, συνετά, χρήσιμα, οικονομικά αποδοτικά και όπως δείχνει το παρελθόν δεν πρόκειται μόνο για την κατασκευή οδών και ξενοδοχειακών αλυσίδων μόνο. Μια πιλωτική φάση, πρώτη φάση είναι πολύ σημαντική γιατί πρέπει να τηρούμε τα υπεσχημένα και αυτή την εποχή έχουν δοθεί πολλές μοιραλιστικές υποσχέσεις σε σχέση με το ομόλογα έργου και μπορεί να δημιουργηθεί σκάνδαλο. Ε, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο δρόμο της αρετής. Ευχαριστώ, κύριος ε, Σον Κέλλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ χάρηκα που μπόρεσα να υποστηρίξω την έκθεση αυτή. Είναι σαφές ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου βρίσκεται από πίσω. Ε, μόνο 32 ήταν κατά και 9 απέσχων. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα. Ε, θέλουμε την πιο στενή συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλους τους εμπλεκομένους. Ε, πρέπει να ε, συμμετέχει και η Ιρλανδία. Εμείς σε θέματα ενεργειακά συνεργαζόμεθα και με το γείτονα το Ηνωμένο Βασίλειο και ελπίζομαι σύντομα και με άλλους. Και σε ό,τι αφορά τις μεταφορές το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σύνδεση με το Eurostar με την υπηρετική Ευρώπη και κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει κάτι παρόμοιο που θα συνδέει την Ιρλανδία με, την, με το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί οι σχέσεις δεν ήταν ποτέ καλύτερες χάρη ιδιαίτερα στην βασίλισσα της Αγγλίας που ε, επισκέφθηκε τη χώρα και την περασμένη εβδομάδα έκανε ιστορική συνάντηση με τον κύριο Μακίνες και ε, νομίζω ότι όλα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στακουλά. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα υποστήριξα την πρόταση και τη βρίσκω πολύ καλή. Είναι σημαντικό τα διευρωπαϊκά δίκτυα να ενισχυθούν οικονομικά και να βρούμε και νέα μέσα. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς θα λειτουργήσουν στην πράξη αυτά τα ομόλογα έργου. Ε, χρειαζόμαστε πάντως έργα καταρχήν που δίνουν ευκαιρίες ανάπτυξης γιατί η ανάπτυξη μας ενδιαφέρει τώρα θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη γιατί το χρέος των χωρών μόνο μέσα από την ανάπτυξη μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ε, υπάρχει ένα καλό έργο λοιπόν που θα συμμετέχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργήσει συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης σε αρμονία με το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος ε, Ντάνιλ Χάναν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μία ακόμα φορά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα. Δηλαδή, υπερβολική κατανάλωση χωρίς παραγωγή είναι η αιτία των προβλημάτων. Ξέρω βεβαίω ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Εάν κανείς πλήξει τους Ευρωπαίους ε, συντηρητικούς, βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να καταλάβουμε το πνεύμα που επικρατεί από άποψη ψυχολογία ενδεχομένως. Ο συνάδελφός μου που είναι ψυχίατρος θα μπορούσε να μας εξηγήσει την έννοια της προβολής. Κανένας ε, βεβαίως ε, δεν χαροποιείται με την κανένα δεν το η οικονομική κρίση. Κανένας, ε, σε κανένα δεν αρέσει να λέει σε, εγώ σας το είχα πει. Δεν γίνεται καθόλου δημοφιλής. Το θέμα είναι να μην κάνουμε διαρκώς τα ίδια λάχη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά που βρισκόμαστε. Δαπανούμε πολλά, ξοδεύουμε πάρα πολλά. Και διαδανειζόμαστε πολλά. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ο τελευταίος ονειδητής. Το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη είναι το ψήφισμα σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Κυρία Πιετικά είναι λόγο. Ευχαριστώ. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και γι' αυτό οι πολιτικές δηλώσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ισορροπημένες. Υποστηρίζω την εξελικτική πορεία και θα πρέπει να εξευρεθεί μια κοινή λύση γιατί υπάρχει μεγάλη ε, ανθρώπινα Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ανθρώπινη τραγωδία και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να σταθεί υπέρ μιας πολιτικής όπου θα σταματήσει αυτή η αδυσόπιτη βία και θα αυξηθεί η ασφάλεια των ανθρώπων στη Μέση Ανατολή. Κυρία Ρομπέρτα Αντζελίλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι κατεπίγουσα η ανάγκη να επιτευχθεί πρόοδο σε ό,τι αφορά την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα το όραμα των λαών τη περιοχή, των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Αυτό είναι καθοριστικό στοιχείο για την ειρήνη και τη σταθερότητα και την ευημερία τη περιοχή. Οι επιθέσει πυράβλων από την ε, ε, Γάζα, οι εκενώσει, η καταστροφή των κατοικιών στην ε, Ιερουσαλήμ, Επιδείνωση των συνθηκών ζωής κυρίως των γυναικών και των παιδιών της Παλαιστίνης. Όλα αυτά είναι παράγοντες που υπονομεύουν την ανέβρεση μιας λύσης. Η λύση, η αντιμετώπιση της σύγκρουσης ε, είναι ένα θέμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Θα πρέπει να απέχουμε από δράσεις οι οποίες διακυβεύουν την αξιοπιστία του σχεδίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη Δυτική Όχθη γίνονται διαρκώς παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό υπονομεύει οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία. Δίνει όθηση στον εθνικισμό και παρακολεί την ανάπτυξη της περιοχής. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας το πρόβλημα των 2.300 Βεδουίνων που υπάρχει περίπτωση να, να εκδιωχθούν από τις ε, κατοικίες τους. Ε, πάρα πολλά παιδιά έχουν αποκλειστεί από την εκπαίδευση το εναλλακτικά μπορούν να πάνε στο ε, Λίβανο, κοντά στην ε, περιοχή της Παλαιστίνης. Αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να σταματήσουν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία κατά της καταπίεσης, κατά της καπάλησης για μια σοσιαλιστική εναλλακτική λύση στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Τάνο. Βρισκόμαστε σε μια φάση ζωτικής σημασίας για την ειρηνευτική διαδικασία και νομίζω ότι εμείς τη στιγμή που ε, έχουμε ταχθεί κατά του Ισραήλ δεν θα πρέπει να παροτρύνουμε για περισσότερες, ε, να εξωθούμε για περισσότερη βία και εντάσεις. Το Ισραήλ ζει σε κατάσταση ευημερίας και δεν είναι σκόπιμο να είμαστε μόνο μονομερείς. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να είναι πιο αντικειμενικό και να μην πιέζει προς εντάσεις οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές δεν υπερψήφισαν το ψήφισμα διότι πρόκειται για μία λιτανία καταδίκης του Ισραήλ ενώ είναι η μόνη δημοκρατική χώρα της ευρύτερης εκείνης περιφέρειας. Θα πρέπει λοιπόν να εξευρεθεί μία ειρηνική λύση. Ο κύριος Στάκουλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταψήφισα την πρόταση, το ψήφισμα αυτό, γιατί ήταν πολύ μονομερές όπως είπαν και άλλοι προλαλήσαντες. Θα πρέπει να θυμούμαστε, θυμούμαστε τις αξίες μας, είμαστε ελεύθερες δημοκρατίες και θα πρέπει να φτάσουμε σε μία ειρηνευτική διαδικασία, να προωθήσουμε την ειρηνευτική διαδικασία και την ειρήνη της ευρύτερης περιοχής η Χαμάς θα πρέπει να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ και να σταματήσει τις επιθέσεις κατά της χώρας αυτής που έχουν ξαναρχίσει πρόσφατα. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τη δημοκρατία, τις αξίες μας και θα πρέπει να πούμε ότι η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ, δεν μπορεί να το μυθι. Και εάν φτάσουμε σε μία διζωνική λύση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, ιστορικά γεγονότα. Ο κύριος ε, Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι θέλουν η ειρηνευτική διαδικασία να παρακολουθηθεί με τρόπο ενεργό. Όλοι ξέρουν επίσης ότι δεν υπάρχει απλή λύση και Όποιος ξέρει την ιστορία και τις εξελίξεις γνωρίζει ότι δεν μπορούμε εύκολα να διαφοροποιήσουμε μεταξύ του καλού και του κακού εκεί. Ως επιτοπλίστων είμαστε στη μέση, στην κρίζα ζώνη. Και βλέπω ότι η πρόταση ψηφίσματος ε, ε, είναι μονοπλευρή γιατί δεν έχουν συμπεριληφθεί τα θεμητά συμφέροντα της Ισραηλινής πλευράς. Είπα, είναι δύσκολο να διακρίνουμε μεταξύ καλού και κακού. Εγώ θα ήθελα μια πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα ήταν ε, ευρύτερη και πιο ισορροπημένη ε, για να συμφωνήσω με την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν ο τελευταίο ομιλητή τη Συνόδου. Έτσι λοιπόν διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τι 3 το απόγευμα. Θα σα δούμε ξανά τότε.